Είναι η έκθεση έγκριτου όσον αφορά την εξωτερική διάσταση τη κοινή ελληνική πολιτική συμπεριλαμβανών και των συμφωνιών αλληλεία. Τώρα για τέσσερα λεπτά θα δώσουμε το λόγο ει την εισηγήτρια. Έχετε το λόγο κυρία Έγκστρομ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, να ευχαριστήσω πρώτα πρώτα όλους τους σκιώδης ηγητές για την ε, καλή συνεργασία που είχαμε. Επίσης και το συμβουλευτικό όργανο το οποίο οργάνωσε την συνάντηση στην Λας Πάλμας και έτσι συνέβαλαν στην ε, σύνταξη αυτής της έκθεσης. Μεγάλη μου χαρά βλέπω ότι όλοι θέλουμε να έχουμε βιώσιμη αλληλεία και ελευτική πόρη να βρίσκονται σε επίπεδο που να έχουμε απόδοση ε, όσο γίνεται μεγαλύτερη αλλά και βιώσιμη και εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι ούτως ώστε να πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί σε σχέση με κάποιες ελευθερικές συμφωνίες γιατί αυτό που θα πρέπει η καινούργια πολιτική να έχει είναι καινούριου ε, κανόνες για το πώς γίνεται η αλληλεία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σεβαστούμε ανθρώπινα δικαιώματα και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα πλεονάσματα. Στην συμφωνία με την Βρετανία ε, συζητήσαμε και θα πρέπει να την εγκρίνει το Κοινοβούλιο και ευχαριστώ κύριε Επιτροπή γιατί γνωρίζω ότι οι διαπραγματεύσεις θα είναι πολύ δύσκολε με την Βρετανία αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να σας πούμε μπράβο γιατί τα πήγατε πάρα πολύ καλά. Τώρα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το ότι θα πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις. Επίσης εμείς θα ε, υποπτεύσουμε την Μαυριτανία να τηρήσει τις δεσμεύσεις της και θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν όλες οι συμφωνίες που κάνουν με ιδιώτες και κρατικούς φορείς. Υπάρχουν πολλά θετικά. Ας πούμε ότι θα, θα υπάρχει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για joint ventures και είπαμε ότι έτσι θα υπάρχει μια πλατφόρμα ε, για να έχουμε βοήθεια πάσης φύσης προς τις ε, τρίτες χώρες. Θα εναρμονίσουμε τις προϋποθέσεις πρόσβασης στα αφρικανικά είδατα για όλους τους ε, στόλους, διαχείριση των αλληλευτικών ε, πόρων, προγράμματα ελέγχου και επίσης ε, θα πρέπει να υπάρξει ένα δίκτυο συμφωνιών ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε και το ότι όλοι και των μακρινών χωρών οι στόλοι θα σέβονται τα συμπεφωνημένα. Άρα θα πρέπει να έχουμε για αυτά τα joint ventures ε, ένα πλαίσιο και να εξασφαλίσουμε το ότι θα είναι αυτές οι κοινέ επιχειρηματικέ δράσεις βιώσιμες. Επίση είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έχουμε κοινού στόχου ε, και έτσι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το ειδικό βάρο μα για να βελτιώσουμε τη διαχείριση των ελληνικών ε, πόρων για να υπάρχει διαφάνεια, να ενθαρρύνουμε επομένω την ε, πρόοδο, να υπάρξει εξουσία προ τα πάνω και όχι προ τα κάτω στην παγκόσμια πολιτική. Ελπίζω ότι η συνεργασία θα διέπεται από θετικό πνεύμα όσον αφορά το νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ είμαι εισηγήτρια στο σχετική έκθεση και από ό,τι ξέρω θα τα συζητήσουμε στην επόμενη σύνοδο. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ο λοιπόν και τρόφιμο διαδικασία Κατσουδιά ελκύω με την προσοχή του Προέδρου. Έχουμε 7 ε, συναδέλφους μου στο λόγο. Πρώτος είναι ο κύριος Μάτο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή που μπόρεσε να στάξει αυτή την καλή έκθεση. Η εξωτερική διάσταση της ε, πολιτικής αλίας είναι σημαντική για την Ευρώπη εάν δούμε την ανεπάρκεια των ε, αποθυμάτων των λευμάτων οι συμφωνίες σύμπραξης είναι ένα... θα έχουν σημαντικό όφελος ε, οικονομικό και κοινωνικό για τους ε, κατοίκους αυτών των ε, ζωνών. Επιπλέον είναι καθαριστικός ο ρόλος στη δημιουργία θέσεων απασχόλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στις χώρες στα των οποίων αλλιεύουν οι Ευρωπαίοι αλείς και μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι ευρωπαϊκοί στόλοι πληρούν ένα υψηλό επίπεδο προδιαγραφών. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και ότι και οι ελευτικοί στόλοι άλλων χωρών πληρούν αντίστοιχες προϋποθέσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος ε, Σάντος. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, για μία ακόμα φορά θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια. Πραγματικά θα ήταν δύσκολο να, να κάνει όλη αυτή τη δουλειά, να πάρει υπόψη της όλες τις ε, διαφορετικές απόψεις των σκιωδών. Έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Μιλάμε για ένα σημαντικό έγγραφο και συμφορώ με τους προλαλήσαντες, όπως ας πούμε τον κύριο Μάτο. Αυτό όμως που δεν επιτεύχθη είναι να δώσουμε την επαρκή σημασία στην θαλάσσια βιοπικιλότητα. Όμως από την άλλη πλευρά υπάρχουν πάρα πολλές πολλά θετικά ζητήματα. Πρέπει να εγκρίνουμε το έγγραφο αυτό. Αναφέρθηκε στον ενιαίο κατάλογο των διεθνών υδάτων γίνεται αλλαγή σημαία αρκετά συχνά και πολλοί ψάχνουν να βρουν την πιο συμφέρουσα. Αυτό είναι μια πρακτική που πρέπει να σταματήσει. Οι που προκαλούνται στον τομέα τη αλληλεία δεν έχουν πλέον εθνοτικά χαρακτηριστικά, καθότι αυτοί που συγκρούονται είναι οι φτωχοποιημένοι από την οικονομική κρίση και τι φορομπηχτικέ πολιτικέ τη λιτότητα αλληλή τη Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία προχωρά στη λήψη μέτρων για την προστασία των θαλασσίων πόρων σε αυτή την κρίση προστίθεται βεβαίως και η διαρκώς αυξανόμενη πίεση που ασκούν οι αναδυόμενες αλλιευτικές δυνάμεις από την ασία καθώς επίσης και η έλλειψη σεβασμού των θεμελιωδών αρχών που η κοινή αλλιευτική πολιτική έχει θεσπίσει. μια εύλογη εξωτερική διάσταση της κοινή αλλιευτικής πολιτικής οφείλει να διασφαλίζει τα συμφέροντα των ευρωπαίων αλλιέων ιδιαίτερα των μικρότερων και να επιτάσσει τη βιωσιμότητα τη διατροφική ασφάλεια και την καταπολέμηση της παράνομης αλληλείας εκτός ευρωπαϊκής ένωσης διότι οι επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα δεν γνωρίζουν όρια. αυτό όμως θα είναι ανώφελο αν η κοινή αλλιευτική πολιτική δεν απαντήσει ταυτόχρονα στο δίκαιο αίτημα ανασυγκρότησης του πρωτογενούς τομέα της ευρώπης ιδιαίτερα σε εκείνες τις χώρες που έχουν πληγεί από τα μνημόνια όπως η ελλάδα. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε τον εισηγητή για την εργασία που επετέλεσε και θα ήθελα να πω ότι ο Ευρωπαϊκός Τόλος η Ευρωπαϊκή επαγγελματίες της, επαγγελματίες είναι σύμφωνη ε, όσον αφορά την ε, εκμετάλλευση των, ε, την εξοπλίση των αποθεμάτων και τις συμφωνίες με τις τρίτες χώρες για την καταπολέμηση της παράνομης ελαθρέας και ανεξέλεγκτης αλίας. Θα πρέπει να ενισχυθούν οι περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλίας, αλλά θα πρέπει ως στόχο να έχουμε μια πολιτική συμπράξεων που να φέρει καλά αποτελέσματα. Ε, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να επωφεληθούν ε, οι δικοί μας ε, λύσει. Ζητώ υπευθυνότητα, σεβασμό και σεβασμό για, έναν, για το κλάδο της αλίας και αυτό είναι το πνεύμα των περισσότερων τροπολογιών που έχουν υποβληθεί σε αυτή την έκθεση. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Φερέρα. εξωτερική διάσταση της κοινής ελευθερικής πολιτικής έχει πολλά μειονεκτήματα, πολλές εσωτερικές αντιφάσεις και γι' αυτό και εμείς ε, έχουμε πάρα πολλά να πούμε κατά αυτής της ισχύουσα σήμερα πολιτικής οπότε υπό την αιγίδα της ε, πολιτικής εταιρικών σχέσεων όλα ε, γίνονται τελικά ε, χρηματοοικονομικές συναλλαγές με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Και έτσι εκμεταλλευόμαστε τους ε, θαλάσσιους πόρους. Μιλάμε για φαινόμενα δεκαετιών. Όμως αυτές οι χώρες έτσι αποστερούνται τις προστιθεμένες αξίες. Θα την είχαν εάν οι ίδιες αυτές οι χώρες εκμεταλλεύονται ε, τους ε, θαλάσσιους πόρους τους. Δεν μπορούν έτσι να αναπτυχθούν, δεν έχουν την κυριαρχία λόγω αυτών των συμφωνιών. Άρα θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχει χρεοκοπήσει η κοινωτική πολιτική σε όλα αυτά και άρα θα πρέπει να γίνουν εκβάθρων αλλαγέ όσον αφορά αυτή την εξωτερική διάσταση τη κοινή ελευθερική πολιτική και να προσέξουν περισσότερο την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Ο κύριο Πόλτσακ, έχει το λόγο, λέει η πρόεδρο. Θα ήθελα, θα να διαπιστώσω ότι η Τσεχία παίρνει χρήματα, κονδύλια από το Ταμείο Αλίας και αυτό, είναι, και αυτό σημαίνει για πρώτη φορά. θεωρώ σημαντικό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολείται με αυτό το ουσιαστικό θέμα, δηλαδή τις αλευτικές συμφωνίες. Στο σημείο 12 αναφέρεται ότι ο βασικός στόχος της ελευτικής πολιτικής ε, ε, θα πρέπει να εγκείται στην αναζήτηση αλευτικών δυνατοτήτων σε τρίτες χώρες. Το Κοινοβούλιο έχει την άποψη όταν ε, οι στόλοι αναλαμβάνουν δραστηριότητες σε τρίτες χώρες θα πρέπει τα αποτελέσματα να ε, τα αποτελέσματα, συγγνώμη, ε, ε, συναρτώνται με άλλα κριτήρια από αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να ασχοληθούμε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πιστεύω ότι οι συμφωνίες σύμπραξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες που συνήθως είναι αναπτυσσόμενες χώρες είναι μεγάλη σημασία και για τις ίδιες τις χώρες γιατί συνήθως έχουν μια επανάπτυκτη αλία ε, μικρής κλίμακας και βιοτεχνική και από, τις, ε, από τα χρήματα τα οποία εμείς ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να επενδύσουμε στις υποδομές εκεί μπορούν να βελτιώσουν τον στόλο τους τόσο στη Μαυριτανία και στο Μαρόκο έχει γίνει κάτι τέτοιο και ε, βάση των κανόνων της κοινή αλευτικής ε, πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό βάσει των ε, επιστημονικών αποτελεσμάτων για τα ηχθειοαποθέματα, είτε αυτό αφορά τον τόνο, στον ειρηνικό ή στην Αφρική, στον Ατλαντικό κλπ. Θεωρώ ότι είναι τελείως σημαντικό να καταπολεμήσουμε την παράνομη αλία και να δούμε ποιες είναι οι χώρες οι οποίες δεν ε, τηρούν τις συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών και αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε καλύτερα όταν οι δικοί μας ελευτικοί στόλοι αναλαμβάνουν δραστηριότητα στα ύδατα αυτών των χωρών. Και νομίζω ότι μπορούμε να συνδυάσουμε τους στόχους αυτούς πολύ καλά με την ε, αναπτυξιακή πολιτική, αυξάνοντας και το επίπεδο ε, το βαθμό της ποιότητας. Και αυτό είναι ιδιαίτερο σημαντικό, γιατί τα ψάρια είναι κοινό αγαθό και ε, υπάρχουν ε, ξεκάθαρες συμβάσεις που μπορούν να επιτηρηθούν με τα διεθνή συστήματα πλοήγησης, ε, γκαλιλαίο κλπ. Ακόμη και τα λεφτικά σκάφη έχουν συστήματα εντοπισμού τους, άρα δεν θεωρώ ότι είναι δικολογημένες τόσες ανησυχίες των συναδέλφων και θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για αυτή την πολύ καλή έκθεση. Ευχαριστώ και τώρα θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο κύριο Βέλα. Thank you, Madam President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί μέλη. Εκτιμώ ιδιαίτερα τη στιγμή κατά την οποία γίνεται η έκθεση αυτή, τη στιγμή που και θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Τις συστάσεις της έκθεσης κινούνται στην κατεύθυνση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου αναγνωρίζει ότι οι βιώσιμες συμφωνίες για την αλληλεία ενισχύουν την ανάπτυξη της αλληλείας στις χώρες εταίρους. Συμφωνώ ότι οι συμφωνίες αυτές παίζουν ένα ρόλο ε, παγκόσμιας διακυβέρνησης των ωκεανών. Όπως γνωρίζετε, στόχος μου είναι να θέσω συγκριτικές, μετρήσεις στο τομέα αυτό. Αυτό αφορά και την ασφάλεια των τροφίμων. Πρέπει να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες να χειριστούν τους, το, τους πόρους με βιώσιμο τρόπο. Και βεβαίως αυτό είναι σημαντικό για την παροχή υγιεινής τροφής και, της, και του βιοπορισμού των ε, παράκτιων κοινοτήτων τα ε ε και συμφωνίες αλληλευτικής σύμπραξης είναι ένας πολύ, είναι ένας, ένα πολύ κατάλληλο εργαλείο για την προώθηση της ε, λογοδοσίας αλλά και της βιωσιμότητας. Συμφωνώ με το στόχο σας επίσης ότι πρέπει να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη συνεκτικότητα μεταξύ της αλληλείας, της εμπορικής και ε, περιβαλλοντικής πολιτικής και της εμπορικής συνεργασίας. Συμφωνώ, όπως επισημαίνει και στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, υπάρχει περιθώριο περαιτέρω βελτίωσης. Αυτό, παραδείγματος χάρη συμβαίνει με την τομεακή πολιτική στήριξή μας που είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο που στηρίζει τους εταίρους των τρίτων χωρών για την πρόθεση αλίας τους με βιώσιμο τρόπο και να αντιμετωπίσουν την παράνομη, αδήλωτη και λαθρεαλία για την εξασφάλιση μεγαλύτερης συνεκτικότητας με τις πολιτικές μας και την περιφερειακή μας συνεργασία. Κάποιες από τις προτάσεις της έκθεσής σας έχουν ήδη συμπεριληφθεί στην πρόσφατη πρότασή μου για την βιώσιμη διαχείριση του εξωτερικού στόλου. Θέλω να βελτιωθεί το ισχύο νομικό πλαίσιο και να διευρυνθεί ώστε να αντιμετωπίζει την κατάσταση, την περίπτωση όπου τα ε, σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλιεύουν ε, εκτός των υδάτων της συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων των ιδιωτικών αδειών όπως ονομάζονται υπάρχουν θέματα που αφορούν σημαίες και που δεν καλύπτονται από τους ισχύοντες κανόνες. Όλα αυτά θα διευκολύνουν τη διαφάνεια και θα αποτελέσουν ένα ακόμα βήμα προς την ενίσχυση της διακυβέρνησης των ωκεανών όπου παίζει σημαντικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσβλέπω λοιπόν στην υποστήριξή σας προς προτάσεις αυτές. Τέλος, δύο λόγια για τις ε, πόδα, τις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλίας. Υπάρχουν ε, ε, περιοχές όπου είναι κοινά τα ευθεία αποθέματα. Έχουμε, συνεργαστεί, έχουμε εργαστεί για να ε, αυξηθεί η απόδοση των πόδα τα τελευταία χρόνια μέσω και επίσης της χρηματοδότησης. Ε, θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την συμμόρφωση με τα επιστημονικά ε, βρήματα και θα, θα τα συμπεριλαμβάνουμε στη λήψη των αποφάσεων. Τα υφιστάμενα συμβουλευτικά σώματα όπως η ε, Αλή, η Επιτροπή Αλίας του Ανατολικού και Κεντρικού Ατλαντικού πρέπει να ε, ε, εργαστούν. Όμως αυτό δεν μπορούμε να το πετύχουμε μόνοι μας. Από την αρχή της θητείας μου προσπάθησα να συνεργαστώ με τους βασικούς παράγοντες για να προωθήσουμε το θέμα. Σε σχέση με το γεγονός ότι η συγκίτρια υποστηρίζει ε, ε, την πρότασή μας για κοινοπραξίες, η Κομισιόν έχει προτείνει συνθήκες για τις νέες προτάσεις της, για τον κανονισμό για τον εξωτερικό στόλο, τον FAR, και ο οποίο είναι υποδιαπραγμάτευση. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνει η διαφάνεια και περιορίζονται οι δυνατότητε κατάχρηση. Με την ευκαιρία αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέλω να σα διαβεβαιώσω, είναι, έχει δεσμευτεί στην πρόθεση της παγκόσμια διακυβέρνηση και τη σημαντική στοιχείου της, της διακυβέρνησης των ωκεανών. Θέλουμε να έχουμε το απαραίτητο νομικό πλαίσιο και διμερός και σε περιφερειακό επίπεδο έτσι ώστε να έχουμε βιώσιμες ε, συμφωνίες αλληλευτικής σύμβραξης για να εξασφαλίσουμε ότι τα αποθέματα θα ε, έχουν την καλύτερη δυνατή διαχείριση με διαφάνεια. Θέλω να ευχαριστήσω το Σώμα για την υποστήριξή του και προσβλέπω στην ε, συνέχιση της, του έργου μας σε πνεύμα συνεργασίας. Ευχαριστώ όλους σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πίτροπε. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Και τώρα, σύμφωνα με την ημερήσια έχουμε τι πανεβάσει διαρκέ ενό λεπτού.